Τον λόγο έχει ο κύριος Μπέγκε για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όντω, συζητάμε σήμερα και πάλι μία πρόταση για να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση ε, διότι οι προθεσμίες μειώνονται συνέχεια και τώρα πρόκειται για αιτήσει από τη Σουηδία και την Αυστρία σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία και από τις κάτω χώρες σχετικά με κατασκευαστικές εταιρείες. Θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν αυτό το ταμείο είχε προβλεφθεί για ε, ένα ότατο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεδομένων των καταστάσεων στο διεθνές ε, πεδίο πρέπει να βασιστεί σε ε, μετεκπαίδευση, σε, σε επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και σε ε, επανένταξη. Γι' αυτό και ε, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, ε, μεμονωμένες ε, εκθέσεις και δεν θα έπρεπε να υπάρχει όπως εδώ για τελευταία φορά ελπίζουμε υπάρχει μια συνολική έκθεση για την κινητοποίηση του ταμείου αυτού και τονίζουμε ότι δεν πρέπει εδώ να αντικατασταθούν τα εθνικά μέτρα ή οι συλλογικές συμβάσεις ή δεν πρέπει να υποκατασταθούν οι δυνατότητες αναδιαρθρώσεως διαφόρων τομέων της οικονομίας. Ελπίζουμε δε ότι συστηματικά οι ε, μεταφορές των πιστώσεων δεν θα γίνονται από το κοινωνικό ταμείο διότι ουσιαστικά το Ταμείο τη Προσαρμογής στην είναι μια ειδική περίπτωση με ειδικέ προθεσμίε. Εδώ έχουμε τρει συγκεκριμένε προτάσεις. Πρόκειται για συνολικά 15,9 εκατομμύρια ευρώ και ε, η ε, Σουηδική και η Ολλανδική πρόταση βασίζονται στο άρθρο 15α για τις ε, απολύσεις δηλαδή πέραν των 500 ατόμων εντός 4 μηνών και η αίτηση της Αυστρίας βασίζεται στο άρθρο 2β δηλαδή τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός 9 μηνών σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επιχειρήσεις και ιδίως μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. Για την Σουηδία πρόκειται για 4.687 απολύσεις στην ε, Volvo και σε 23 προμηθευτές της και ζητούσε η ε, Σουηδία 9.839.000 ευρώ. Η αίτηση της Αυστρίας ε, αναφέρεται στην επιχείρηση Steiermark και υπευλήθη στην Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 2009 για 744 πωλήσει και για ένα ποσό 5.705.000 και η αίτηση των κάτω χωρών υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Αυγούστου 2009 αφορά 570 πωλήσει και ε, ζητούν 386.114 ευρώ. Ε, θεωρούμε ότι τα κριτήρια καλύπτονται από τις αιτήσει αυτές για να ικανοποιηθούν και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Απασχολήσεως σύμφωνα με την διαδικασία έχει επίσης ε, ε, καταρτήσει μία γνωμοδότηση πολύ προσεκτική ιδίω στην περίπτωση της Σουηδίας διευκρινίζει ότι από τις 4.600 απολύσεις εδώ αναφερόμαστε μόνο σε 1.500 επίσης ότι στην Heymans υπάρχουν επίσης επιπλέον 400 απολύσεις από συμβασιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση δηλαδή υπάρχει μία σειρά περιπτώσεων η οποία εδώ δεν πρέπει να μας εμποδίσει να χορηγήσουμε εξετάσουμε τις άδειε αυτές. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σπίτλα, κύριε Πίτρο, έχει το λόγο. Βάζενη Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο στόχος της πρότασης αυτής είναι η κινητοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο λόγω των απολύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Σουηδία, την Αυστρία αλλά και στην κατασκευαστική βιομηχανία στις κατοχώρες. Ο εισηγητής ε, εκφράζει την υποστήριξή του μαζί με κάποιες ε, προτάσεις σχετικά με τον προπολογισμό, τις οποίες είχα τη δυνατότητα να συζητήσω και σε προηγούμενες ευκαιρίε. Θα επανέλθω. Το πρώτο σημείο που αφορά τον προπολογισμό έχει να κάνει με τι πηγές χρηματοδότηση. Μα υπενθυμίσατε ότι δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι το μόνο που χρηματοδοτεί. Το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα δημοσιονομικό ειδικό εργαλείο το οποίο δεν έχει ίδιου πόρου αυτό καθεαυτό. Επομένω, για να γίνει η κινητοποίησή του θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πιστώσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, βρούμε τις κατάλληλες ε, πιστώσεις ε, και η αρχή θα, επί του προπολογισμού αρμόδια θα πρέπει να απελευθερώσει, να αποδεσμεύσει με τροποποίηση του προπολογισμού τα κονδύλια αυτά. Και αυτό γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίε προκύπτουν. Είναι γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέχρι στιγμή ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότηση. Και αυτό όχι μόνο διότι ομοιάζει με άλλες πηγές χρηματοδότηση. Έχει δηλαδή σημαντικά κονδύλια. Ένα δις περίπου ευρώ το 2009 σε ό,τι αφορά πιστώσεις ε, πληρωμών. Από αυτό το ποσό τα 6 χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές ε, προς το Ευρωπαϊκό Τομείο την Παγκοσμιοποίηση, ήταν 53 εκατομμύρια το 2009, δηλαδή 0,5 κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μέχρι στιγμής ε, η μέθοδος που έχουμε ακολουθήσει, μια μέθοδος που φαίνεται να είναι εύλογη αλλά και βολική, δεν έχει καθυστερήσει ούτε όμως θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ωστόσο, συμφωνώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στις πηγές πληρωμών. Σας διαβεβαιώνω ότι από πλευρά Επιτροπή δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και ελπίζω στο μέλλον να είμαστε σε θέση να σα παρουσιάσουμε περισσότερε επιλογέ. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέτεται δεν αφορά μόνο τον προπολογισμό, αλλά και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσει για την κινητοποίηση του Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση σε ξεχωριστά έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα πλεονεκτήματα μια τέτοια διαδικασία. Παραδείγματο χάρη, θα εξαλείψει τον κίνδυνο μυστικών συμφωνιών. Είναι γεγονό ότι η πρωτότυπη αρχική μέθοδο που χρησιμοποιούμε φαίνεται να είναι η φυσική οδός που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Διότι καθιστά ευκολότερη τη διαχείριση. Αν όμως δείτε την ουσία και τις πολιτικές πτυχές, φαίνεται ότι αυτές μας οδηγούν σε μια διαδικασία κατά περίπτωση. Αυτό το οποίο προτίθεται και η Κομισιόν να πράξει από εδώ και πέρα. Αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος ε, Φανίστεροι για δύο λεπτά. Voorzitter, ongewone tijden vragen om ongewone maatregelen. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τα μέτρα που προτείνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης είναι πολύ συγκεκριμένα. Κατά τρόπο ώστε τα λόγια να μεταφερθούν και να μεταφραστούν σε πράξεις. Τα προτινόμενα μέτρα που αφορούν τις κατασκευαστικές εταιρείες και το μεγάλο αριθμό απολύσεων εκεί και για τη δική μας χώρα αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέτρα σημαντικά. διότι ακριβώς οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία μας. Οι δράσεις που θα πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδευτούν από την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης είναι πολλοί αυτοί που έχουν βρεθεί σε μειονεκτική θέση Αλλά μιλάμε εδώ για εργαζομένους με συγκεκριμένε δεξιότητες που μετά από λίγα χρόνια θα μας λείψουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν τις δεξιότητες αυτές, τις ικανότητες των εργαζομένων να τις ε, προφυλάξουμε και οι περιφερειακές μα αρχέ και οι αρχές του Μπραμπάντε θέλουν να επενδύσουν σε δράσεις για τη στηρίξη των υποδομών και του τομέα αυτού και εσωτερικά και εξωτερικά στη χώρα. Είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και μόλις την τελευταία εβδομάδα στα πλαίσια της Συνόδου της Κοπενχάγης συζητήθηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά με την ενέργεια, προκειμένου να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και των μεταφορικών μέσων. Εδώ μιλάω και για τα περιφερειακά ταμεία, τα οποία θα πρέπει να επιταχύνουν τη δράση τους και να την συγκεκριμενοποιήσουν. Ελπίζω το Κοινοβούλιο λοιπόν να στηρίξει όλες αυτές τις ιδέες. Θα πρέπει να στοχεύουμε την ποιότητα και την διάρκεια. Οι τρεις, λοιπόν αυτές οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι ιδιαίτερα εύστοχες και τις στηρίζω.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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κινητοποίηση αυτού του ταμείου ζητάται όλο και περισσότερο και αυτό οφείλεται στην ε, οικονομική κρίση ε, η οποία μαστίζει την Ήπειρό μας. Ε, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις τελευταίες τρεις αιτήσει για την αυτοκινητοβιομηχανία και την κατασκευαστική εταιρεία οι οποίες έχουν γίνει δεκτές θετικά. Πρέπει να να σας πω ότι ε, πλέον ε, έχει προσθεθεί ε, το χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε θετικά τις αιτήσει. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε καλύτερα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τους πολίτες μας και βλέπουμε από την την έκθεση του κυρίου Μπόγκε γιατί ότι χρειάζεται να υπάρχει μία επιτάχυνση ε, της διεκπαιρεώσεως και να, να βρεθούν και άλλα ταμεία πέραν του κοινωνικού ταμείου. Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να υπάρξουν πλήρες πιστώσεις πληρωμών αλλά γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου επ' αυτού του θέματος και ε, παρακολούθησα τα σχόλια του Επιτρόπου. Βεβαίως υπάρχει καλή θέληση και ελπίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του Ταμείου θα μπορέσει να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους στόχους, τους μας και να ενισχύσουμε αυτό το Ταμείο. Thank President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή εκδήλωση αλληλεγγύη προ του εργαζομένου που έχουν χάσει τι δουλειέ του λόγω σημαντικών δομικών αναδιαρθρώσεων. Ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να αισθανόμαστε κάποια ικανοποίηση με το ότι μπορούμε και εμεί να συνεισφέρουμε στην ελάφρυνση ορισμένων άμεσων ε, επιπτώσεων των απολύσεων για τους εργαζόμενους και να τους δώσουμε δηλαδή κάποια ελπίδα για το μέλλον. Ωστόσο, δεν θα πρέπει απλά να βελτιώσουμε αυτό το ταμείο. Έχουμε ευθύνη να κάνουμε πάνω το δυνατό ώστε να εξασφαλίσουμε πρώτον ότι ε, πληρούνται όλα τα κριτήρια, αλλά και να κάνουμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση να δώσει προστιθέμενη αξία ένα από τα συναφή ζητήματα που έχει θέσει και η Επιτροπή Απασχόληση είναι ότι τα προτινόμενα από τα κράτη-μέλη μέτρα συμπληρώνουν άλλε δράσει συγχρηματοδοτούμενε από τα διαδοτικά ταμεία. Και πραγματικά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από την απλή επιβεβαίωση ότι περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να αποδειχθεί, να καταδειχθεί ότι περί αυτού πρόκειται, γιατί αυτό θα βοηθήσει να βρεθεί αυτή η προστιθέμενη αξία για την οποία μίλησα. Επίση, η προστιθέμενη αξία θα προέρχεται από το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν θα αντικαθιστά δράσεις που είναι ευθύνη εταιριών, αλλά θα προσθέσει μέτρα σε αυτά τα οποία λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και όταν αξιολογήσουμε την προσθέμενη αξία ε, για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο ε, της αναθεώρησης του πολιτικού προγράμματος, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καθιερώσουμε ως πάγια τακτική και να, είμαστε, να επαγρυπνούμε. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κοιτάζοντας την κατανομή αναφύλως, στα τρία αυτά προγράμματα για την παροχή βοήθειας, βλέπουμε ότι 91, 72 και 79% είναι άνδρες αυτά ε, τα άτομα. Και έχω δει και άλλα προγράμματα που έχουμε χρηματοδοτήσει. Φαίνεται να υπάρχει μία ε, ένδειξη ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης προς άρενες ε, απολυθέντες εργαζομένους. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μια στατιστική επεξεργασία για τον ένα ή τον άλλο λόγο να είναι αυτά τα νούμερα έτσι. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ προσεκτικά όλε τι αιτήσει. γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει ενίσχυση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Η κυρία Κορνελίσεν για δύο λεπτά. Laat ik vooropstellen dat wij Αυτά τα προτινόμενα μέτρα τη Επιτροπή Απασχόρτη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και τι τρει προτάσει που έχουμε στα χέρια μα, Πιστεύουμε ότι τα κονδύλια θα φτάσουν στα χέρια των ενδιαφερόμενων δικαιούχων. Όμω, το πλαίσια του Ταμείου αυτού υπάρχει μια σημαντική έλλειψη. Διότι αυτή τη στιγμή αποδεχόμαστε να βλέπουμε και να θεωρούμε την ε, ευρωπαϊκή οικονομική αγορά με μια πολύ συγκεκριμένη θεώρηση για το μέλλον. Όμως δεν είμαι βέβαιη ότι έχουμε καθορίσει μια συγκεκριμένη πορεία για το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο διορατική προσέγγιση και πιο μακροπρόθεσμη. Υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσης θα πρέπει να προβλέψουμε τέτοια επιτόκια που να μας επιτρέψουν να ανακάμψει η οικονομία μας κατά τρόπο βιώσιμο. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό το ταμείο μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, αλλά σίγουρα είναι ένα εργαλείο. Όμως δεν δίνει οριστικές λύσεις. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, κάποιες γενικές κατευθύνσεις ώστε οι πολίτε να μην κοιτάζουν μόνο το παρελθόν προ τα πίσω για να αισθανθούν καλά, αλλά να μπορούν να κοιτάζουν με αισιοδοξία και το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε συγκεκριμένε κατευθύνσει για μια οικονομία που να επιτρέπει σε όλου να ωφεληθούν. Ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι. Εδώ γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εάν θα έπρεπε να σταλούν προς την Σουηδία, τις κάτω χώρες ή την Αυστρία που έχουν ζητήσει να ενισχυθούν για τις απολύσεις οι οποίες έχουν γίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε μία κατασκευαστική. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες ερωτήσεις και στο παρελθόν, αλλά δεν είναι σωστό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει αυτό το σκεπτικό γιατί δεν είναι δίκαιο. Οι πιέσει των ανταγωνιστών ε, επηρεάζουν όλους τους εργαζομένους και όλους τους εργοδότες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο κάθε μέρα εξαφανίζονται πολλές θέσεις εργασίας αλλά δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας και μια τέτοια ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται μόνο σε μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός απολύσεων. Οι μικροί εργοδότες όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέτρο αυτό άρα το μέτρο είναι επιλεκτικό και άδικο. Δεύτερο επιχείρημα πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να επιλύονται σε εθνικό επίπεδο διότι οι πόροι υπάρχουν και μπορούν να διατεθούν εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τους απολυμμένους εργαζομένους στην Σουηδία, την Αυστρία και την Ολλανδία. Όμως, κάθε αίτηση για κινητοποίηση του ταμείου αυτού ουσιαστικά μας οδηγεί σε, περισσότερους, σε περισσότερες απορίες για το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό και δίκαιο. Για την αποτελεσματικότητά του, ήδη το 2009 πρέπει να πούμε ότι το Ταμείο αυτό στήριξε 16.000 εργαζομένου. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των απολυμμένων εργαζομένων. Ε, τώρα μιλάμε για στήριξη τριών εκατομμυρίων στι εκατοντάδε εκατομμύρια που μπορεί να βρεθούν χωρί ε, δουλειά. Πού είναι η δικαιοσύνη λοιπόν. Ε, στηρίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία με 500 εκατομμύρια και 314 για τον αυστριακό τομέα τη ίδια βιομηχανία. Ενώ στην Πορτογαλία Έχουμε 524 εκατομμύρια στήριξη μόνον και στην, Καταλα... στην Καταλωνία μπορεί να λάβουν βοήθεια 2.000 εκατομμυρίων. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για εκπρόθεσμες αιτήσει και πώς θα βρούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι που σωστά ωφελήθηκαν από το Ταμείο. Εδώ θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τη διακριτική μεταχείριση στην ε, ανεργία και την καταπολέμηση της έλλειψης ισορροπής μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων χωρών. Ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει δημοσιονομικά μέτρα για να στηρίξει τους εργαζομένους που βρίσκονται χωρίς δουλειά λόγω των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο εμπορικό σύστημα παγκοσμίω και πολλέ από αυτέ έχουν προκληθεί από πρωτοβουλίε έμεσε ή άμεσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, εδώ στόχο είναι να επιδοτήσουμε και την εκπαίδευση αυτών που έχουν χάσει τη ε, δουλειά του, αλλά δεν θα επιλύσουμε έτσι τα προβλήματα τη ανάλογη βιομηχανία. Ούτε θα δημιουργήσουμε εναλλακτικού τομεί βιομηχανία που θα προσφέρουν υπηρεσίε και θέσει εργασία για αυτού του εργαζομένου. Εδώ σπαταλάμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι είναι μέρο τη κρίση που προκλήθηκε και να ε, διερευνήσει τα αίτια για τις κρίσεις Θα πρέπει να μην ενεργούμε ως φιλάνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν τους φτωχότερους. Βεβαίως, οι δράσεις αυτές αρχικά θα ανακουφίσουν, θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες τους, τους πολίτες της μάλλον. Αλλά η έκθεση και η έτσι ψηφίσματο όπω ε, προτείνονται για ψηφοφορία δεν καταδεικνύουν ποιο θα, είναι, ποιο θα είναι το πεδίο των χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή πόσε βιομηχανίε θα καλύπτονται και πόσε εταιρείε ε, σε κάθε βιομηχανικό κλάδο. Αυτό που είναι πιο ενισχυτικό όμω είναι ότι η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι πληρωμέ μέσω των επιδοτήσεων, χωρί όμω να αποτούνται αποδεκτικά στοιχεία ότι τα κονδύλια φτάνουν στου σωστού δικαιούχου για το σωστό σκοπό. Πρέπει εδώ να απαιτήσουμε τακτική παρακολούθηση των προορισμών των χρηματοδοτήσεων και τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων βάσει τη διαδικασία του 2007-2013 και του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Συνάδελφοι, εδώ μιλούμε για χρήματα των φορολογουμένων. Πολλοί από αυτού έχουν ήδη χάσει τη δουλειά του ή δεν παίρνουν καμία επιδότηση, καμία στήριξη. Πολλοί από αυτού ζουν δυσμενεί οικονομικέ ε, στιγμέ. Πώ λοιπόν θα ωφεληθούν από αυτά τα χρήματα. Εγώ απορρίπτω το ψήφισμα αυτό και σα καλώ να κάνετε το ίδιο. Κύριε Βέρθμαν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση έχει ένα δημοσιονομικό μέτρο που μπορεί να βοηθήσει οικονομικά τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη διεθνή κρίση. Και αυτό ισχύει και για την δικιά μου περιοχή η οποία έχει πληγεί. Έχω πει ότι το, το Ταμείο της παγκοσμιοποίησης δεν πρέπει να παρανοηθεί, πρέπει να εξυπηρετεί κατευθείαν τους πολίτες και γι' αυτό θα πρέπει να ελέγχεται και θα ήθελα να, υπάρχουν, να υπάρχει παρακολούθηση και ε, μία αναφορά σχετικά με την πρόοδο χρηματοδότησης της Steiermark η οποία είναι ένα θετικό παράδειγμα για την χρήση των ε, οικονομικών πόρων υπέρ των πολιτών. Ε, για λεπτά.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 Ευχαριστώ κύριε και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι γιατί συζητάμε σήμερα για το πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν φταίνε και δεν έχουν τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν την, την οικονομική κρίση και ε, δεν έχουν οικονομικούς πόρους ε, χαιρετίζω λοιπόν τη γέφυρα αυτή η οποία καταρτίζεται με τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν επιχειρήσεις αυτές ε, την χρηματοδότηση προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Πρέπει να αναλύσουμε ε, ακριβώς πού έχουμε πραγματικά βοηθήσει να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίες και πού καταφέραμε να ε, εντάξουμε και πάλι τους απολυμένους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας και να τους βοηθήσουμε άμεσα. Πρέπει να βοηθήσουμε άμεσα γι' αυτό και θα πρέπει η κινητοποίηση να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ιδίω στην αυστριακή περίοδο, ε, στην αυστριακή περιοχή, στην ε, Steiermark, όπου πρόκειται για μια κατασκευαστική εταιρεία η οποία είναι πολύ σημαντική και για τον χώρο της. Είναι καλό να μπορέσουν να διατεθούν αυτά τα 5,7 εκατομμύρια. Θα πρότεινα όμως σε όλες τις περιπτώσεις να τις αξιολογήσουμε θετικά και να γίνει μία ανάλυση. Όχι απλώς να ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα, αλλά να μπορούν να δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις, να υπάρξει μία ενεργή οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή η οποία θα ενισχυθεί ε, σχέση με ό,τι υπήρξε στο παρελθόν και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. η αίτηση της Αυστρίας για στήριξη από το Ταμείο Προσαρμοποίηση αναφέρεται εις ε, ε, ε, επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία ή στην περιοχή της Στηρίας, στην Στάιερμαρκ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή και μπορεί να βοηθήσει και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση διότι αν χαθούν οι θέσεις εργασίας ε, μπορεί ε, να αντισταθμίσει την ανευθυνότητα των χρηματαγορών διότι ε, υπάρχουν πολλές επιπτώσεις της κατάρρευσης της ζητήσεως στην αυτοκινητοβιομηχανία που επηρεάζουν μία περιοχή ιδίω όταν πρόκειται πρόκειται για φορτηγά. Βλέπουμε εδώ ότι μειώθηκε σχεδόν κατά 60% η ζήτηση ε, φορτηγών και αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή η επένδυση είναι εξαιρετική για να μπορέσουν να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίες τα, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι. Δηλαδή θα μπορέσουν τα 5.705.000 ευρώ να χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιηθούν ε, για να μπορέσουν ε, να, ε, να εφαρμοστούν μέτρα επαγγελματικού προσανατολισμού. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κάπνοχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα υποτίθεται θα σχολιάζαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την κινητοποίηση κεφαλαίων ε, για τρεις περιπτώσεις, Αυστρία, Σουηδία, κάτω χώρες από το Ευρωπαϊκό Τομείο Υποστήριξη Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Παρ' όλα αυτά, οι τρει αυτέ περιπτώσει ε, είναι τελείω διαφορετικές η μία από την άλλη και δεν σχετίζονται μεταξύ του. Θα σα υπενθυμίσω ότι έχει γίνει στο παρελθόν όταν είχαμε ζητήσει ε, από την ε, Κομισιόν να μα κάνει ξεχωριστά, να μα παρέσει ξεχωριστά αυτές τις προτάσεις. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ασαφ... πολλές ασάφειες στις προτάσεις αυτές. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε πόσα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την Σουηδία. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αυστρία, το ποσό Πραγματικά είναι εντυπωσιακό για τον κάθε απολυθέντα. Ήταν εκατοντάδες ευρώ, αλλά τώρα ζητά πάνω από 14.000 ε, για τον κάθε απολυθέντα η Αυστρία και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό συμβαδίζει με την ε, πρόταση για το Ταμείο. Δεν θα υποστηρίξουμε λοιπόν την κινητοποίηση του Ταμείου. Ο κύριος Ρούμπιξ σήκωσε μπλε κάρτα. Το επιτρέπετε? Ναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την μπλε κάρτα απλώς για να διορθώσω. Δεν δίνεται η βοήθεια αυτή μόνο για ένα άτομο στην Αυστρία. Πρέπει να διορθώσω. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπετε προφανώς ότι είναι ένα αυστριακό θέμα και η Στηρία είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ αφενός από την κατάρρευση της αυτοκινητοβιομηχανίας και ιδίως ε, ε, από την κατάρρευση της εξαγωγικής δραστηριότητας διότι ε, ε, υπήρξαν όπως ε, λέχθη ένας πολύ μεγάλος αριθμός απολύσεων οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν 744 ουσιαστικά θα έπρεπε όμως να διευκρινίσουμε σε σχέση με τον προλαλήσαντα ότι δεν πρόκειται απλώς για επιδοτήσεις για αναδιάρθρωση αλλά για στήριξη των εργαζομένων με ε, μέτρα επανακπαίδευσης, με οικονομική στήριξη άμεση διότι όπως ελέγχθη πρέπει να μπορέσουν να προβούν σε επαγγελματικό αναπροσανατολισμό για να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους, να αποκτήσουν ε, νέες δεξιότητες όπως παραδείγματο χάρη στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Ο επόμενος είναι ο κύριος Χάρμαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε μια τέτοια συζήτηση είναι σημαντικό να θυμίζει κανείς ότι η παγκοσμιοποίηση είναι και αυτό που έκανε εύπορη την Ευρώπη. Μας έφερε ευημερία, θέσεις εργασίας, επενδύσεις, εξαγωγές. Αυτό μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε νέες εταιρείε, οι οποίες έγιναν και πολυεθνικές, εισαγωγής ε, και εισαγωγές γενικότερα, έδωσαν άλλες ευκαιρίες στους πολίτες μας να έχουν ποιοτικά προϊόντα, ποιοτικές υπηρεσίες σε καλές τιμές. Αυτό λοιπόν αφορά μια ολόκληρη γενιά και μιλάμε για αλλαγέ ευρύτατης κλίμακας, οι οποίες συνεχίζουν να εκτελήσονται με νέες εταιρείε, με νέες ε, υπηρεσίες που προσφέρονται. Αυτά συνεχώς αναδύονται. Τώρα, οι σημερινές συνθήκε ε, πλήττουν ολόκληρη την κοινωνία και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τις αναχαιτίζουμε απλώς. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να διευκολύνουμε να συμβούν να δώσουμε νέες δυνατότητες στα κράτη-μέλη ώστε ε, να γίνουν οι αλλαγέ και να προσαρμοστούμε σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Για το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα, προφανώς δεν μπορεί να δώσει ίσε ευκαιρίε σε όλους ή όπως άλλα υποθετικά μέτρα θα μπορούσαν. Θα ήταν παραπλανητικό να πούμε ότι τα πράγματα θα ήταν ε, απλό να επιληθούν μόνο μέσω του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήταν ε, θαυματουργό ένα τέτοιο μέσο. Α σκεφτούμε την αυτοκινητοβιομηχανία στην Αυστρία. Ε, υπάρχουν πολλές συνεισφορές από όλη την Ευρώπη και θα μπορούσαν να γίνουν χρηματοδοτήσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις εθνικές αρχές. Όμως το πρόβλημα είναι και η στρέβλωση του ανταγωνισμού. ιδίω όταν μιλάμε για κρατικά κονδύλια τα οποία παρέχονται σε ένα βιομηχανικό κλάδο συγκεκριμένο. Αυτό θα ήταν στρέβλωση. Ή μια άλλου είδου στρέβλωση θα ήταν να δημιουργήσουν να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα σε εταιρείε που δεν είχαν ίσε ευκαιρίε για χρηματοδότηση σε άλλε επαρχίε τη χώρα, σε άλλε χώρε. Παρόλα αυτά είμαστε υπέρ τη πρόταση, διότι τώρα αυτή η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Οι συνεισφορέ αυτέ μπορούν να καταβληθούν και είναι πολύ αργά για να γυρίσουμε τώρα πίσω και να παρακάμψουμε τι στρεβλώσει. Ευχαριστώ. Η επόμενη είναι η κυρία Μωράν Σαρτιέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αποβλέπει εις την βελτίωση των δυνατοτήτων απασχολησιμότητος των εργαζομένων. Εκεί πρέπει να επέμβουμε και έτσι πρέπει να καταρτήσουμε τους φακέλους τους οποίους ε, καταρτίζουμε για το Ταμείο Προσαρμογής για να μπορέσουν να διατηρηθούν στην αγορά εργασίας δεν υπάρχει ένταξη κοινωνική χωρίς επαγγελματική. Επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά και θα ήθελα να ζητήσω από τις αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες πλήττονται από αυτή την κρίση να προσαρμόσουν τις προσφορές τους εις ε, τις επιταγές του περιβάλλοντος και στις ανάγκες των καταναλωτών για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αλλά ευχαριστώ τον κύριο Μπέγκε για την πρότασή του και θα ήθελα όπως το έκανε και ο κύριος Ρούμπικ να ε, παρακολουθήσουμε ότι η πολιτική μας εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Τίκαου με τη διαδικασία Catch the Eye. Πέρσι εγκρίναμε πολλές, πολλά μέτρα στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Κοσμοποίηση προκειμένου να διευκολύνουμε τους εργαζομένους που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω των αλλαγών στη δομή του παγκόσμιου εμπορίου. Η κρίση έπληξε τι υποδομέ του διεθνού εμπορίου και παρατηρήσαμε το 2009 είχαμε τουλάχιστον 2.500 απολύσεις στη Χαλιβουργία και 700.000 στις κατασκευαστικές εταιρείες. και στον σιδηροδρομικό τομέα εξίσου. Είναι λοιπόν σημαντικό το 2010 να είμαστε προετοιμασμένοι για, μεγάλες, για μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Λόγω ακριβώ αυτών των οικονομικών αλλαγών θα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι και η διαδικασία διάθεση των κοπηλίων να είναι πολύ απλή, ώστε οι δικαιούχοι και τα κράτη να έχουν ε, πρόσβαση στο Ταμείο. Η Σουηδία, η Αυστρία και οι κάτω χώρε έχουν καταθέσει την αίτησή του ήδη από τον Ιούλιο. Οι κάτω χώρε, μάλλον πιο συγκεκριμένα τον Αύγουστο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μια και βρίσκομαι εδώ και ακούω αυτή τη συζήτηση και μιλάμε για το Ταμείο, Παγκοσμιοποίησης, Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, πρέπει να πω ότι πολλοί εργαζόμενοι απολύθηκαν διότι η εταιρεία στην εκλογική μου περιφέρεια συγκεκριμένα μετακίνησε εργοστάσια της στην Πολωνία τα μέτρα που προτείνονται σήμερα για την Αυστρία, τη Σουηδία και τι κάτω χώρε ε, έτυχαν πολλών σχολείων. Εδώ το θέμα είναι πρέπει να σκεφτούμε τι ποσά θα προβλέψουμε, για ποια διάρκεια και πώς θέλουμε να τα ταπανίσουμε. Όχι μόνο για δύο χρόνια πρέπει να παράσχουμε στήριξη, αλλά πρέπει να στηρίξουμε και τις υποδομές. Και θα πρέπει οι κυβερνητικοί φορεί να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και να παράσχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους επιχειρηματίες. Το 35% των νέων εταιριών στην Ευρώπη ε, τελικά ανήκουν σε ιδιοκτήτες που έχουν μείνει χωρίς εργασία. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η ένδυα έχει γίνει μια σύγχρονη εφεύρεση και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι ομιλητοί στη διαδικασία Catch the Eye. Α, και νομίζω το λόγο έχει τώρα η Επιτροπή. Όχι, βλέπω κάποιον ακόμη. Εάν θεωρήσουμε ότι περισσότερες ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη οφείλονται ε, στην παγκοσμιοποίηση και γι' αυτό κινδυνεύουν, θα πρέπει να προσέξουμε οι νέοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θεωρούνται καν άνεργοι γιατί δεν έχουν ε, τελειώσει ακόμη τις σπουδέ τους ή την επιμόρφωσή τους να βοηθηθούν. Και ιδίως στην Αυστρία θα έπρεπε οι εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας να στηριχθούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν με πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενταχθούν στην ε, αγορά εργασίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρξει κάποιος άλλος ο οποίος ζητά το λόγο και θα δώσω και πάλι το λόγο στον Επίτροπο Σπίτλα. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πολύ καλή και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έγιναν πολλές αιτήσει και το Ταμείο έχει χρησιμοποιηθεί προς όφελος των τελικών δικαιούχων. Ως Επίτροπος πάντοτε προσπαθώ να εξετάζω τα αποτελέσματα επιτόπου και να αποκτώ άμεση γνώση των θεμάτων. Έτσι λοιπόν εκτίμησα ε, και εγώ ε, την θετική αξιολόγηση πάντοτε του Ταμείου και των αποτελεσμάτων του. Η συζήτηση έδειξε βέβαια ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο επί παραδείγματι, το γεγονός ότι το Ταμείο είναι χρήσιμο μόνο για μεγάλες εταιρείες. Ευτυχώς η πρακτική έχει δείξει ότι ο αρχικός σκοπός που ήταν η χρησιμοποίηση του Ταμείου για όλα τα κρατη και για όλα τα είδη εταιριών και μεγεθών εταιριών τελικά ε, αποδίδει υπάρχουν κανόνες που μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό και για υπαλλήλου μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από την κρίση και αυτό χωρίς καμία διάκριση. Θα ήθελα να τονίσω το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ταμείου. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει άτομα και όχι εταιρείες δεν μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύουμε το Ταμείο αυτό ως ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να βοηθά μη βιώσιμες εταιρείε. Όχι. Το αντίθετο ισχύει. Το Ταμείο αυτό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει άτομα που έχουν απολυθεί και να τα βοηθήσει συγκεκριμένα να βρουν γρήγορα και εύκολα μία νέα θέση εργασίας. Είναι ένα ταμείο λοιπόν που μας βοηθά να προωθήσουμε την αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω ποιος το είπε, νομίζω ήταν η κυρία Χάρκιν, ε, η οποία εξέφρασε την ε, ανησυχία της ε, για πιθανή μη ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Ναι, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία υπάρχει αυτή η ανισότητα, αν θέλετε, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι η κρίση έπληξε τομείς ε, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι άρενες, δηλαδή κατασκευές, ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Σε, αυτές, ε, σε αυτούς τους κλάδους απασχολούνται κυρίως άνδρες. Εξού έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι περισσότερη υποστήριξη δόθηκε σε άρενες εργαζομένους. Ο πρόεδρος Ομπάμα μάλιστα είπε ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ Πολιτειών είναι, θα είναι γυναίκες. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά έχουν πληγεί τυπικά ανδροκρατούμενοι ε, τομείς ε, οικονομική δραστηριότητα, εξού και βλέπετε αυτή την ανισότητα. Επίσης ακούσαμε στη συζήτηση πολλές ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί το Ταμείο κάτι το οποίο είναι άθικτο, απαραβίαστο, δεν κανείς δεν πρέπει να το αγγίξει, είναι ταμπού ή οτιδήποτε. Φυσικά και μπορεί να υποστεί αλλαγές και μεταβολές. Δεν υπάρχει επί της ουσίας κάποιο εμπόδιο. Ένα άλλο ερώτημα, ένα άλλο ζήτημα είχε να κάνει με τον τρόπο της χρηματοδότησης. Ότι δηλαδή θα πρέπει να πράξει μια ξεχωριστή γραμμή, ένα ξεχωριστό κονδύλιο προπολογισμού. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών που ισχύουν δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο παρότι συζητήθηκε σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι κινητοποίησαμε τα κονδύλια αποτελεσματικά αλλά με άλλο τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ναι πράγματι Λόγω της πίεσης από την κρίση θα υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, περιπτώσεις τέτοιες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της όλα τα επιχειρήματα τα οποία λένε ότι πάντοτε θα πρέπει να ακολουθούμε κατά περίπτωση διαδικασία και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και στο μέλλον. Θα εξετάζουμε δηλαδή την κάθε περίπτωση χωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Προεπολογισμών και όλους τους βουλευτές ε, που ε, έδειξαν ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα. Διότι πράγματι η συζήτηση έδειξε ότι εξετάστηκαν όλες οι πιθανές ε, πτυχές σε σχέση με αυτό το ταμείο. και ε, αντίστοιχε τέτοιε περιπτώσει είναι επιλέξιμες και θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμε και στο μέλλον αντίστοιχε περιπτώσει για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτή η συζήτηση λοιπόν έδειξε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή και ελπίζω να είναι θετική και η ψήφος των Ευρωβουλευτών. Ε, Ευχαριστώ ε, τον κύριο Πίτροπο και για να κλείσει τη ζήτηση έχει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε ο Επίτροπος. Συμφωνώ μαζί του, ιδίως όταν στο τέλος αναφέρθηκε στη μελλοντική χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ε, ιδίως σε σχέση με άλλα ταμεία όπως το κοινωνικό, επί του οποίου θα έχουμε μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για τους εργαζομένους. Δεν είναι αυτός ο στόχος του, αλλά μπορεί να βοηθήσει με μονομένα ε, περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και που μπορούν να προβούν σε μια αναδιάρθρωση επαγγελματική και ε, να αλλάξουν πορεία. Και βεβαίως ε, βάσει της επικουρικότητας μπορεί να βοηθήσει συμπληρωματικά το Ταμείο ταμείο αυτό το κοινωνικό ταμείο το οποίο διαθέτουμε και θα ήθελα να σας πω ότι βεβαίως θα πρέπει να αμφισβητούμε περισσότερο ε, την αποτελεσματικότητα άλλων ταμείων και όχι τόσο αυτού νου το οποίο ε, προσπαθεί να βοηθήσει συγκεκριμένα άτομα. Ευχαριστώ. Λίγη συζήτηση αυτή και θα, η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Η κυρία Μπερέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημειώνω ότι σε όλη την προηγούμενη συζήτηση λέγατε ότι θα υπάρξει τώρα